Επιτροπή σχετικά με τον απολογισμό της Δανικής Προεδρίας και θέλω να χαιρετήσω την απερχόμενη εκπρόσωπο της ε, Προεδρίας της Δανίας και της ε, δίνω τον λόγο. Εδώ είναι σήμερα και ο Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, κύριος Μπαρόζο και ξεκινάμε κατευθείαν με τη συζήτηση και τον πρώτο λόγο έχει η Πρωθυπουργός της Δανίας κυρία Τόνι Σμιτ Έχετε το λόγο κυρία μου. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμη ε, πρόεδρε των πολιτικών ομάδων, κύριοι ευρωβουλευτές, ε, κυρίες μου. Είναι μεγάλη τιμή μου να απευθύνομαι